Señorías, reanudamos la sesión. En primer lugar, he de hacer dos anuncios. El primero es que... Καλησπέρα σα. Ας αρχίσει η συνεδρίαση. Ε, ο κύριος Σιγνάτη παρετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 23 Απριλίου και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού μας ε, λαμβάνουμε γνώση της απουσίας του από την ημερομηνία αυτή και μετά και θα ενημερώσουμε και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Δεύτερη ανακοίνωση. Στην συνάντηση του Απριλίου η Νομική Επιτροπή ενέκρινε την διαπίστευση των συναδέλφων Μπαουτίστα και Λίπινων. Και επίσης προτάθηκε με ομόφωνη γνώμη όλων την έγκριση της εντολής τους. Και αν δεν έχετε κάποια ένσταση θα θεωρήσω ότι η απόφαση αυτή έχει επικυρωθεί και τώρα. Σύμφωνα με τη μερισσία διάταξη προχωρούμε στην ε, συζήτηση εκθέσεως Κρόλη που αφορά τη διάρκεια προστασία του δικαιώματο της πνευματικής διοκτησίας μένων συγγενικών δικαιωμάτων. Πρώτα πρώτα ο κύριος συζητή έχει το λόγο, ο κύριο Κρόουλη για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε κύριο Μακρύβη στην αίθουσα και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που βρίσκονται μαζί μα. Αυτή η παρέκταση τη προστασία του δικαιώματο αποτελεί κάτι πολύ το